Chers collègues, j'aimerais vous inviter à prendre place parce que... Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Πρέπει να επιδείξουμε τεράστια πειθαρχία ε, για να συγκροτηθούν σε σώμα σήμερα όλες οι επιτροπές που έχουν προγραμματιστεί. Για το λόγο αυτό λοιπόν, μετά από μια μικρή ανάσα που θα πάρουμε, θα ε, προεδρεύσω τη συνεδρία σας. Καλωσορίσατε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι στη συνεδρίαση συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού μας προεδρεύω προσωρινά μέχρι να εκλεγεί πρόεδρος ε, στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους και όλες. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ε, οπότε θα πρότεινα να αρχίσουμε αμέσω. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης. Θυμίζω ότι μοναδικό αντικείμενό μας είναι η συγκρότηση σε σώμα με εκλογή Προέδρου και τεσσάρων αντιπροέδρων σύμφωνα με το άρθρο 213 του Κανονισμού Λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχάς, θα εκλέξουμε Πρόεδρο και στη συνέχεια έναν έναν τους τέσσερις αντιπροέδρους θα σας ε, ανακοινώσω τα ονόματα των αναπληρωματικών που συμμετέχουν στην ψηφοφορία και θυμίζω ότι θα πρέπει να ε, με ενημερώσουν πριν αρχίσει η ψηφοφορία οι πολιτικές ομάδες αν έχει αλλάξει κάτι ως προς τα ονόματα. Αναπληρωματικά μέλη λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο κύριος Λούκας Μάντελ αντικαθίσταται από τη Μαρλένε Βόχτλερ και η Γιαννίνα Πογιώσκα από την κυρία Εύα Κόπατς. Καλά τα είπα. Καλά τα καταγρεώργησα τα ονόματα των δύο αναπληρωτών, αλλά πρόκειται για τα πρόσωπα αυτά που αντικαθιστούν ε, τα τακτικά μέλη. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Λοιπόν, οι σοσιαλιστές και δημοκράτες δεν έχουν ανακοινώσει αναπληρωματικά μέλη. Ρινιού. Ο κύριος Μάρτιν Κόγουτ αντικαθίσταται από την Μαρία Σοράγια Ροτρίγκες Ράμος. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σχετικά. Για τις λοιπές πολιτικές ομάδες της Επιτροπής μας δεν έχω τίποτα νεότερο. Η ομάδα ID, η ομάδα ECR, η Ενατική Αριστερά και η μία εγγεγραμμένη έχουν ονόματα αναπληρωτών να ανακοινώσουν. Εν τη αυτή περίπτωση, προχωρούμε στην εκλογή του Πρόεδρου μας. Απαρτία έχουμε. Παρίσταται το 1 τέταρτο των μελών μας. Επτά βουλευτές, μόνο επτά, πολλούς περισσότερους. Παρακαλώ, ε, υποψηφιότητες για την Προεδρία. Θα ήταν κρίμα να μην έχουμε κανένα πρόεδρο. Θα προτείνει κάποιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ως ε, νέα συντονιστή, ε, συντονιστής θα ήθελα να προτείνω τον κύριο Τόμας Τόμπεϊ ως πρόεδρο. Ε, το σημειώνω Άλλη υποψηφιότητα έχουμε. Θυμίζω ότι οι υποψηφιότητες θα πρέπει να κατατεθούν είτε από μια πολιτική ομάδα είτε από ένα εικοστό των μελών της Επιτροπής, δηλαδή δύο βουλευτές στην περίπτωσή μας. Διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα. Comme il n'y δεδομένου ότι έχουμε ένα και μοναδικό υποψήφιο, συμφωνείτε με την υποψηφιότητα αυτή διαβοής. Εάν δεν ρωτήσαμε αν συμφωνεί ο υποψήφιος, υποθέτω ότι συμφωνεί η σιωπή του προς απάντησή μας. Il a Α, συμφώνησε. Θυμίζω ότι θα πρέπει να είναι τακτικά μέλη υποψήφοι, πράγμα που ισχύει, και να έχουν ε, υπογράψει, συμπληρώσει τη δήλωση που θα Okay. Je vous Έλεγα λοιπόν, yes, συμφωνεί ο υποψήφιος. Ah, Θυμίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είναι τακτικά μέλη της Επιτροπής υποψήφοι και να έχουν συμπληρώσει ε, κανονικά τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων, καθώς επίσης και ε, τη δήλωση για τον κώδικα δεοντολογίας. Κύριε Τόμα Τόμπεϊ, σας ερωτώ, ε, έχετε πληρώσει αυτά τα προαπαιτούμενα. Μάλιστα. Καλά, δεν αφέβαλα ούτε στιγμή. αλλά το επιβεβαιώνετε κι εσείς. Οπότε, επειδή δεν υπάρχει παρά ένας υποψήφιος, προτείνω να σας εκλέξουμε διαβοής remake γιατί το ξανακάναμε προηγουμένως. Κάντε λίγη φασαρία για τον πρόεδρό μα. Je constate que vous avez été élu par des applaudissements. Ήταν ε, πραγματικά εκοφαντικό το χειροκρότημα ε, και προαπαιτούμενα για ε, την εκλογή σας. Συγχαρητήρια. Και εγώ ταπεινά αποχωρώ. Thank uh, uh, uh, Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Μεγάλη μου τιμή η εκλογή μου ως πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης. Ε, είδατε πόση λαχτάρα είχα. Είχα ανέβει πριν ε, εκλεγώ ε, επίσημα. Πραγματικά θέλω να σας γνωρίσω όλους στην Επιτροπή. Προσβλέπω σε αυτό. Γνωρίζω ότι στην Επιτροπή Ανάπτυξης έχετε εξαιρετικό μητρό ε, διακομματική συνεργασίας και θα ήθελα να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση. Έχουμε πάρα πολλά σημαντικά θέματα να κάνουμε που μας περιμένουν. Χονδρικά ε, μας αναλογούν 50 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι τα τρία τέταρτα του συνόλου ε, προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική δράση. Έχουμε και τις διαπραγματεύσεις για την εποχή μετά τη Συμφωνία του Κοτονού. Ε, έχουμε να ορίσουμε νέους επιτρόπους. Και στο τέλος της περίοδου αυτής θα είμαστε έξι χρόνια ε, ε, μόλις πριν την υλοποίηση της Ατζέντας για το 2030 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ξέρω ότι γίνεται μέγας λόγος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ποια είναι η σημαντικότερη επιτροπή. Για μένα είναι το ΤΙΔΟ. Sure elected Και ε, όλα τα μέλη της Επιτροπής μας πραγματικά πιστεύω ότι είναι προσιλωμένα και αφοσιωμένα στα θέματα της ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ και πάλι για την εμπιστοσύνη. Πραγματικά προσβλέπω στη συνεργασία μας. Αλλά ας προχωρήσουμε ε, και στις υπόλοιπες εκλογές που έχουμε, που είναι εκλογή πρώτου αντιπροέδρου πρώτα. Με το σημείο 2 δηλαδή στην ημερήσια διάταξή μας. Και σας θυμίζω τα ονόματα των αναπληρωτών που θα συμμετέχουν στην εκλογή των αντιπροέδρων. From EPP, ε, Από το ΕΛΚ, Μαρλέν replacing Lucas Mandel. And we will have Eva Kopacz replacing Janina Okcha. And from Renew, we will have Maria Soraya Rodriguez Ramos replacing Martin Horwood. Okay? Perfect. So if there are no changes to the list, then... Αν δεν υπάρχουν αλλαγές σε αυτά τα ονόματα που σας ανέγνωσα, θα σας παρακαλούσα να κάνετε τις προτάσεις σας ε, για τη θέση του πρώτου αντιπρόεδρου. Μία-μία οι προτάσεις. Alors, ε, προτείνω εγώ, λέει η κυρία Ρίβαζη. Πρώτα ένα σούπερ αντιπρόεδρο. Μία. Πιερέτε Μπερξέ φωνα Σήκω να συστηθεί βεβαίω. Και ε, που κάνει διδακτορικό στην ε, γαλλόφωνη ε, λογοτεχνία έχει συστήσει μία μήκυο κατά του ακροτηρισμού των γενικείων ε, γεννητικών οργάνων και στη Γερμανία εκπροσωπεί τις γυναίκες αφρικανικής καταγωγής ε, για την έρευνα και την ανάπτυξη. Είναι πραγματικά μια πολύ αξιόλογη συνάδελφος νεοεκλεγήσα και μπορούμε διαβοής να την εκλέξουμε. Thank you so much. are there any... Ευχαριστώ πολύ. Άλλες προτάσεις. Θαυμάσια. Ε. Συμφωνείτε με την υποψηφιότητά σας. Πιερέτ. Yes, perfect, perfect. Uh, now we're not there yet. I was also early before, you know. Εντάξει, ακόμα δεν έχουμε βρει το βηματισμό μας και εγώ νωρίς σηκώθηκα. Θυμίζω ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής μας και να έχει ε, συμπληρώσει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων και ε, το κώδικα διοντολογίας. Πληρείτε αυτά τα τρία προαπαιτούμενα, μάλιστα. Θαυμάσια. Ωραία, λοιπόν. Δεδομένου ότι έχουμε μία υποψηφιότητα και μόνο για την πρώτη αντιπροεδρία, προτείνω να την εγκρίνουμε διαβοής, να την εκλέξουμε μάλλον. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας ως πρώτη αντιπρόεδρος της Επιτροπής και σας παρακαλώ να έρθετε εδώ να ε, καταλάβετε τη θέση σας στο Προεδρείο. So, there seems to Λοιπόν, δεν φαίνεται να υπάρχουν ε, αλλαγές. Συνεχίζουμε για τον, ε, την εκλογή του Δευτέρου Αντιπροέδρου. Thank you very much. Ε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για την δική σας εκλογή και για την εκλογή της πρώτης Αντιπροέδρου εξ, ονόματος, συγγνώμη, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών σας ευχαριστούμε για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Ελπίζουμε να είμαστε όλοι μια καλή ομάδα. Θα ήθελα να προτείνω τον κύριο Νόιζα, τον Όρμπερτ Νόιζα. Είναι παλαιό μέλος αυτής της Επιτροπής από την αρχή που βρέθηκε στο Κοινοβούλιο αποφάσισε να είναι ένας από τους ανθρώπους που ασχολείται με τα θέματα της ανάπτυξης, ήταν συντονιστής μας και έχει τεράστια πείρα. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Νόιζα αν συμφωνεί να... για την πρόταση αυτή. Να σας θυμίσω ότι θα πρέπει να είστε πλήρες μέλος της Επιτροπής, θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει πλήρως την δήλωση οικονομικών συμφερόντων και ε, την συμφωνία σας ε, με τον κώδικα συμπεριφοράς. Συμφωνείτε? Ναι, συμφωνώ, λέει ο Νόιζα. Συνεπώς, μιας και υπάρχει ένας υποψήφιος για τη θέση του Δευτέρου Αντιπροέδρου, Προτείνω να εκλέξουμε τον Νόμπερτ Λόιζε για διαβοής. Ε, congratulations on your election as... Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Ελάτε παρακαλώ στο Προεδρείο. Περνάμε στην εκλογή του τρίτου αντιπροέδρου. Να σας θυμίσω, αν υπάρχουν αλλαγές στον κατάλογο των αναπληρωτών, θα πρέπει να μας το γνωστοποιήσετε πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Λοιπόν, ε, υπάρχει πρόταση για το διορισμό του τρίτου αντιπρόεδρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ομάδα Renew Europe προτείνει την κυρία Ζαχαροπούλου, είναι Ελληνίδα, εκλέγεται στη Γαλλία στα πλαίσια του ψηφοδελτίου του Πρόεδρου Μακρό. Έχει πάρει δίπλωμα από το Ιταλικό Πανεπιστήμιο της Σαπιέντσα, είναι γυναικολόγος, έχει κάνει διδακτορικό στα θέματα της ενδομητρίωσης έχει ξεκινήσει μια εθνική εκστρατεία στη Γαλλία για την ευαισθητοποίηση ε, της κοινωνίας στο πρόβλημα αυτό και έχει εκπροσωπήσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρμόδιες επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών. Και γενικά συμμετέχει στις προσπάθειες αυτονόμησης οικονομικής των γυναικών και της πλήρους συμμετοχής τους την οικονομία και την αγορά εργασίας. Λοιπόν, ε, συνοπτικά τα είπα, υπάρχουν πολύ περισσότερα. Perfect. Uh, thank you so much. Σας ευχαριστώ. There seems to be no other nomination, but then I ask... Δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Η κυρία Ζαχαροπούλου, συμφωνείτε με την πρόταση. Ναι, λέει η κυρία Ζαχαροπούλου, να σας υπενθυμίσω ότι θα πρέπει να είστε πλήρες μέλος της Επιτροπής, θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει πλήρως την δήλωση για τα οικονομικά συμφέροντα και τον κώδικα συμπεριφοράς να τον έχετε προσυπογράψει. Ναι, λέει η κυρία Ζαχαροπούλου και στα τρία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, εφόσον είστε η μόνη υποψηφία για τη θέση του τρίτου αντιπροέδρου, προτείνω την εκλογή σας διαβοής.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 Να σας θυμίσω ότι όταν υπάρξει αλλαγή στους υποψηφίους που θα μπουν στην ε, ψηφοφορία για τον τρίτο αντιπρόεδρο θα πρέπει να μας τους κοινοποιήσετε πριν ε, ξεκινήσει η διαδικασία εκλογής. Να ε, δούμε τώρα τις υποψηφιότητες για την εκλογή του τετάρτου αντιπρόεδρου. Πολύ ε, νέος Γερμανός Ευρωβουλευτής εργάζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό με τους νέους πράσινους στην Ευρώπη. Είναι φωτογράφος και φωτορεπόρτερ εδώ και ε, μερικά χρόνια και συμμετείχε σε ε, πολλές ε, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο. Με διάφορες μεταναστευτικές οδούς ακολουθώντας από το Βαλκάνι έφτασα και μέχρι το Αφγανιστάν. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επικεντρωθεί στις πολιτικές μετανάστευσης, το άσυλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά δικαιώματα που είναι και αντικείμενα όλα αυτά της Επιτροπής μας πεπισμένη ότι θα διακριθεί εδώ στην Επιτροπή. Ο κύριος Έρικ Μάρκαρτ. Σήκω. Uh, Ωραία. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια άλλη υποψηφιότητα. Συμφωνείτε για την υποψηφιότητά σας. Συμφωνώ λέει ο κύριο Φάρχαρτ. Λοιπόν, η... πρέπει να είσαστε, να σα θυμίσω, πλήρω μέλο τη Επιτροπή. Πρέπει να έχετε συμπληρώσει τη δήλωση των οικονομικών συμφερόντων και αυτή του ε, κώδικα. Πληρείτε και τα τρία αυτά κριτήρια. Ναι. Ωραία. Οπότε, εφόσον υπάρχει μόνο ένα υποψήφιο για τη θέση του τετάρτου αντιπροέδρου τη Επιτροπή Ανάπτυξη, προτείνω να εκλέξουμε διαβοή. Congratulations Συγχαρητήρια λοιπόν για την εκλογή σας ως τετάρτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας. Παρακαλώ, ελάτε να πάρετε τη θέση σας. Ωραία. Αφού λοιπόν ε, εκλέξαμε τους τέσσερις αντιπρόεδρους, να πω ότι το γλωσσικό καθεστώ της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης είναι αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ουγγρικά, ιταλικά, λιθουανικά, πολωνικά, ισπανικά και σουηδικά. Τώρα, Πάμε στην ε, επιβεβαίωση του ημερολογίου για τα ραντεβού μα για τις συνεδριάσεις μας για το 2019. Έχετε ήδη λάβει το ημερολόγιο, το έχουμε στείλει ηλεκτρονικός μαζί με την πρόσκληση για τις επόμενες συνεδριάσεις. Συμφωνείτε να επιβεβαιώσουμε αυτές τις ημερομηνίε για τις συνεδριάσεις μας. Αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις, τότε επιβεβαιώνουμε και το, ε, τις συνεδριάσεις μας και να σας πω ότι ε, έχει διανεμηθεί και το ε, πακέτο καλωσορίσματος στους ε, νεοεκλεγέντες. Περιλαμβάνει πολύ σημαντικές πληροφορίες για τη δουλειά που κάνει η Επιτροπή μας και τις βασικές της προτεραιότητες. Ωραία. Πάμε στο σημείο 7, επόμενη συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής θα γίνει εδώ στις Βρυξέλλες, στις 23 Ιουλίου του 2019 από τις 5 μέχρι τις 6.30 θα γίνει κοινή μεικτή ε, συνεδρίαση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος για να υπάρξει ενημέρωση για το, ε, υψηλό, για το ε, φόρουμ του υψηλού, υψηλού επίπεδου που θα γίνει αυτή τη βδομάδα και την επόμενη στη Νέα Υόρκη. Η πλατφόρμα επίση του ΟΗΕ, η κεντρική πλατφόρμα για, την, για το θεματολόγιο για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη, για του οποίου θα ενημερωθούμε. Έχουμε λοιπόν σημαντικά θέματα επ' αυτού. Εμεί δεν έχουμε ε, αντιπροσωπεία να στείλουμε εκεί, οπότε είναι σημαντικό να λάβουμε τι σχετικέ πληροφορίε. Επόμενη συνάντηση 24 Ιουλίου από τις 9 μέχρι τις 12.30 και Σας ευχαριστώ πολύ όλους, ευχαριστώ συνάδελφοι, συγχαρητήρια και πάλι για την εκλογή όλων σας. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στην Επιτροπή και να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία βεβαίως που προετοίμασε. Α, συγγνώμη, με συγχωρείτε, παρακαλώ. Ε, κανονικά πρέπει να έχουμε και τα διάφορα στην ημερήσια διάταξη, αλλά εντάξει. Ε, μπορούμε να έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου. Πρέπει να οργανωθούμε και να είμαστε ενημερωμένοι θα μπορούσε κάποιος να μας ανακοινώσει ανεπίσημα έστω το τι θα ακολουθήσει. Ξέρουμε ότι υπάρχει διάσκεψη στη Νέα Υόρκη για την αηφόρο ανάπτυξη, αυτό το ξέρουμε, αλλά υπάρχουν φαντάζομαι και άλλες αποστολές, άλλα θέματα, άλλες αντιπροσωπείες και ίσως πρέπει να είμαστε ενήμεροι. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Οι πληροφορίες που έχω αυτή τη στιγμή είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα πάει η αντιπροσωπεία μας στη Νέα Υόρκη, 23 με 26 Σεπτεμβρίου θα γίνει η συνεδρίαση. Θα είναι παρόντες και τα μέλη της ε, Επιτροπής Ανάπτυξης και τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος. 15 μέλη θα έχει η αντιπροσωπεία αλλά να το ελέγξω καλύτερα με τη γραμματεία και βεβαίως μετά μόλις έχουμε τις ε, πληροφορίες θα σας τις ε, στείλουμε έτσι ώστε να ε, μπορέσετε κι εσείς να προγραμματίσετε τις δραστηριότητε σας. Εντάξει. Και οι συντονιστές επίσης θα έχουν την δυνατότητα να συναντηθούν και να συζητήσουν για τις διάφορες αποστολές, αλλά ακόμα προφανώς δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ακόμα τώρα γίνονται οι εκλογές. Κοιτάξτε, είμαστε μια μικρή επιτροπή. Καλό θα είναι να κυκλοφορούν οι πληροφορίες, έστω και αν επίσημα. Γιατί αν το παίζουμε πολύ επίσημη, θα ναι. καθυστερήσουμε. Φυσικά, όπως σας είπα, θα σας διαβεβαιώ ότι θα ενημερωθείτε. Είμαστε μια μικρή επιτροπή.